Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τρόφιμα τα οποία είναι απολύτω βρόσιμα. Είναι απολύτω ανόητο σε οικονομικό επίπεδο. Είναι σαν να πετούσαμε χαρτονομίσματα στον σκουπιδοντενεκέ. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Έχω πάρει από το Συμβούλιο τις θέσεις που έχουν εγκριθεί από τη, στην πρώτη ανάγνωση ε, και ε, έχουν γίνει δεκτά. Ε, επομένως, οι τίτλοι θα ε, διομοσιευθούν στα πρακτικά της επόμενης Ολομέλειας. Η προθεσμία υποβολής αντίθεσης λίγη αύριο. Επίσης, σας λέγω ότι το ΕΛΚ έχει υποβάλει τα ε, ακόλουθα αιτήματα. Ο κύριος Αντώνιο Καντσάν, μέλος της Αντιπροσωπείας για σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο, θα αντικαταστήσει ο κύριο Αλφρέντο Αντωνιώτσι. Ο κύριος Αλφρέντο Αντωνιώτσι ε, θα, θα αντικαταστήσει τον κύριο Καντσάν στην ε, κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Κροατίας. Επίσης, ο κύριος Ανδρέα Κατσολίνα θα γίνει μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών μετά από αίτημα των Σοσιαλιστών. Κύριε έχετε κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Κανείς λοιπόν δεν αντίθεται στις προτάσεις ε, αυτές. Τα πρακτικά της ε, παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν στην έκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επόμενη συνεδρίαση. Αν ε, δεν έχει κανείς αντίρρηση, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της σήμερα θα μεταδοθούν ως ήθιστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κέλλη, ευχαριστώ εις το μόνο σας ευχαριστώ πάρα πολύ.